Ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτς. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ για την λήψη φωτογραφιών. Ο κύριος Μπροκ μάλλον. Ο κύριος Έλμαρ Μπροκ προεδρεύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρο για την, ε, ιδιαίτερα για την σημερινή συνεδρίαση και θεωρώ ιδιαίτερη τιμή μου που έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Φερκόφνα Ράντα καθώς και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σχεδόν το ίδιο μεγάλη χαρά μας και για την παρουσία εδώ του Επιτρόπου Χάν καθώς και του φίλου Πατ Κόξ που επετέλεσε σημαντικό έργο για λογαριασμό μας σε σχέση με την Ουκρανία και που εξακολουθεί να επιτελεί σημαντικό έργο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ όλες και όλοι που ήλθατε είτε από την Ουκρανία είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, βλέπω και τον κύριο Τουρμπίνσκι και νομίζω ότι η αντίληψη που έχουμε αναπτύξει στην ομάδα στήριξης για την δημοκρατία και συντονισμό των εκλογών ειδικώ για τη συνεργασία με την Ουκρανία και που είναι ένα πραγματικό πρόγραμμα συνεργασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντική και θα υπενθυμίσω με την ευκαιρία αυτή δύο γεγονότα. Όταν κυρώθηκε η συμφωνία συνεργασίας έγινε εκ παραλίλου κύριοι Σούλτς και Γκρόισμαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Φερχόφνα Ράντα την Ουκρανική Βουλή και στην βάση συμφωνίας που έχετε συνυπογράψει και οι δύο. Ο δε συνάδελφός μου, ο Ευρωβουλευτής κ. Πλένκοβιτς, ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, έχει αναλάβει τη σχετική εργασία και χαίρομαι επίσης, όπως είπα, ότι ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δραστηριοποιείται, κ. Πατ Κόξ δηλαδή, πάλι στο πλαίσιο αυτό. Επιθυμούμε συνεργασία η οποία θα διασφαλίσει αμοιβαία τις δυνατότητες μεταρρυθμίσεων και από τις δύο πλευρές με αμοιβαία στήριξη βασισμένη στις εμπειρίες μας για την ε, επανεπεξεργασία κοινοβουλευτικών μεθόδων, την ε, στήριξη της σταθερότητας ε, του Κοινοβουλίου. Σας έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας όπως έχετε και εσείς τα δικά σας, αλλά είναι σημαντικό στα κρίσιμα θέματα να υπάρχει συνεργασία. Γι' αυτό και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα μπορέσουμε να συζητήσουμε διεξοδικότερα τα θέματα αυτά και ιδίως το πόση σημασία αποδίδουμε στις μεταρρυθμίσεις που έχετε αναλάβει στο χώρο της κρατικής δομής, της καταπολέμησης της διαφθοράς, στα θέματα των συνταγματικών αναθεωρήσεων, για την ανάπτυξη από πλευρά της ικανότητας πρόκλησης αυτών των μεταρρυθμίσεων ώστε να μην δοθεί αλωθεί στην άλλη πλευρά για να εμποδίσει την λήψη κάποιων αποφάσεων. Διότι και αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί επειδή δεν υπήρχαν σχετικέ συμφωνίες. Αυτά θα μπορέσουν να συζητηθούν σε ομάδες εργασίας. Χαίρομαι διότι ήδη η συνεργασία αποδίδει καρπούς ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο δηλαδή μια ανεξάρτητη Ουκρανική Δημοκρατία βασισμένη στο κράτος δικαίου στις αρχές της οικονομίας της αγοράς και θέλω και από τη δική μου σκοπιά του Προέδρου δηλαδή της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι, να δηλώσω ότι είμαστε αποφασισμένοι να σας υποστηρίξουμε απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική στάση της Ρωσίας και ότι θεωρούμε ότι όσο η συμφωνία του Μίνσκ δεν εφαρμόζεται, δεν επιτρέπεται να αρθούν οι κυρώσεις. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον ε, συνάδελφο Πλένκοβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε Μπρόκ, αξιότιμε πρόεδρε Σούλτς, αξιότιμε πρόεδρε της Βέχοβνα κύριε Γκρόσμαν, κύριε Πίτρο Πεχάν, ε, κύριε Κόξ, κύριε και κύριοι. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση ω Ευρωβουλευτή και μάλιστα αρμόδιο για την εφαρμογή του προγράμματος θεσμικής αρρωγής και ανάπτυξης ικανοτήτων της Ουκρανικής Βουλής της Βέρχοβνα Ράντα να ε, συμμετέχω εδώ στην ε, επίσημη τελετή έναρξη τη εβδομάδα τη Ουκρανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα είμαι επικεφαλή και τη αντιπροσωπεία για τι σχέσει με τη Βέρχοβνα Ράντα και ε, μέλος της Επιτροπής ε, για την Διακοινοβουλευτική, της τη Επιτροπής ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης. Και κάθε εβδομάδα για μας είναι εβδομάδα της Ουκρανίας. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη εβδομάδα. Και αυτό το λέω ως φίλος και ως συνάδελφος που θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας για να σας βοηθήσουμε, να σας συνδράμουμε ώστε με ειρηνικό τρόπο να ανακτήσετε τα κατεχόμενα και την παράνομα, να ανακτήσετε την παράνομα προσερτημένη Κρυμαία, να εξομαλύνετε την κατάσταση στον Τονέτς και να εφαρμόσετε την Συμφωνία Σύνδεσης ε, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη βοήθεια της αντιπροσωπείας μας και χάρη και στην συνεργασία με τον πρέσβη τον Μπίνσκι. Είναι εξαιρετική και ιδιαίτερα αξιόλογη η έκθεση του κυρίου Κόξ που εκπώνησε μαζί με εμπειρογνώμονε και στο οποίο συμμετείχαν πολύ σημαντικοί θεσμικοί παράγοντες που εδώ και χρόνια βοηθούν τη Βίρχοβνα να ανακτήσει το δυναμικό και τις ικανότητές της και θα αποτελέσει σημαντικό εγχειρίδιο και οδηγός για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στη Βερχοβναράντα και θα συμβάλλουν στην ευημερία όχι μόνο της Ουκρανικής Βουλής αλλά του συνόλου του Ουκρανικού λαού και θα προετοιμάσει το κοινοβούλιο σα να ετοιμαστεί για την μελλοντική φάση και σύνδεσης ε, και προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν ένα χρόνο και τέσσερις ε, μήνες ανέλαβα το έργο και μάλιστα είχα προτείνει τη διοργάνωση αυτής της εβδομάδας της Ουκρανίας ε, στον κύριο Σούλτς και στον συμπρόεδρο Μπροκ. Έγινε ε, επιτέλους ε, έλαβε σάρκα και οστά αυτή η πρόταση και ε, θα συνυπογραφούν και συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των γραμματιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βέρχοβνα Ράντα Και σας εύχομαι πολύ επικοδομητικό και καρποφόρο έργο αυτή, αυτό το τρίμερο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος Μάρτιν Σούλτς. Σας ευχαριστώ και σας κύριε Πρόκ και σας κύριε Πλένκοβιτς. Πρώτα πρώτα ένα θερμό καλώ ορίσατε στον φίλο μου Βλάντιμιρ Γκρόισμαν, πρόεδρο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως ε, το καλώ ορίσατε και για όλες και όλους ε, τους συναδέλφους μας από αυτήν την ε, Ουκρανική Βουλή. Καλώς ορίσατε και εσείς κύριε Χάν, καθώς ένα θερμό καλώς ορίσατε και για τον προκάτοχό μου στην Προεδρία της Ευρωβουλής, κύριο Πατ Κόξ. Έχω εδώ μια ομιλία που δεν θα την εκφωνήσω όμως, διότι όσα είχα γράψει στην ομιλία μου τα είπαν ήδη οι δύο συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα. Είμαι, ε, ε, συνήθως οι ομιλίες μου είναι εφιούς χαρακτήρα, όμως τα είπαν τόσο ωραία που θα αρκεστώ να δείξω στο πόσο ευφύης ήταν δικές τους παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, πάντως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γράφεται κοινοβουλευτική ιστορία. Τα όσα συμφώνησε και τα πράγματα επί των οποίων συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Ουκρανικό δεν έχουν υπάρξει ποτέ, δεν έχουν προηγούμενο. Και δεν μιλώ μόνο για την κοινή κύρωση την οποία επιτύχαμε με χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών, ώστε να την υπογράψουμε ταυτόχρονα, μιλώ και για τις προγραμματικές κατευθύνσεις της συνεργασίας μας σε ό,τι αφορά την ουσία, που θεωρώ ότι είναι υποδηματικές. Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες επιδράσεις έχουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις από άλλα κοινοβούλια τα οποία εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μας με τον ίδιο τρόπο όπως το Ουκρανικό διότι προκαλείται το ενδιαφέρον άλλων βουλευτών που έρχονται και με ρωτούν δεν μπορούμε να κάνουμε μια παρόμοια συνεργασία όπως κάνετε με την Ουκρανία. Αυτό δείχνει ότι στην δημοκρατική συνεργασία, στη συνεργασία προς ένα εκδημοκρατισμό μπορούν, ναι, μπορούμε να ακολουθήσουμε και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την πάρα πάρα πολύ συναρπαστική οδό. Θα ήθελα να απευθύνω το λόγο τώρα και σε όλους τους συναδέλφους μου από εθνικά κοινοβούλια, καθώς και τους ευρωβουλευτές, διότι θεωρώ ότι μαζί με τους συναδέλφους μας του Κοινοβουλίου του Κιέβου γνωρίζουμε και οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ταραχώδης η καιρή και στην Ουκρανία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και την εργασία και τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου του Κίεβου και κάθε φορά που σας βλέπω αγαπητές συνάδελφες στην οθόνη σκέπτομαι τι θαυμάσια δουλειά που κάνω διότι πάντοτε σκεπτόμουν ότι η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια πολύ περίπλοκη υπόθεση, αλλά θαυμάζω και βγάζω το καπέλο μου πραγματικά στο συνάδελφό μου, διότι είναι πολύ πιο περίπλοκη η δική του δουλειά, του Πρόεδρου του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Η συνεργασία μας πάντως συνεχίζεται, η εργασία στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο συνεχίζεται και χρειαζόμαστε σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Χρειαζόμαστε μια σταθερή Ουκρανία. Αντιμετωπίζουμε άνευ προηγουμένου προκλήσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άμεση γειτονία μας ζει δραματικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές μας υποχρώσεις ως Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ζούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση μια κρίση αλληλεγγύης. Το προσφυγικό που αντιμετωπίζουμε μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα στη βάση της αλληλεγγύης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η βασική αρχή της αλληλεγγύης και αυτό πρέπει να ισχύει και προς τα μέσα και προς τα έξω, ως δράση δηλαδή προς τα έξω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προηγουμένη εβδομάδα δέχθηκα εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον πρόεδρο του Λιβανικού Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου του Λιβάνου. Ο Λίβανος με 4 εκατομμύρια, με 4 εκατομμύρια κατοίκους έχει υποδεχθεί 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. σχεδόν 30% των ανθρώπων που διαβιούν σήμερα στον Λίβανο είναι πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμφωνήσει αν θα δεχτεί εν τέλει ένα εκατομμύριο πρόσφυγες για να τους διανύμει ανάμεσα στους 500 εκατομμύρια κατοίκους των 28 χωρών μελών. Γι' αυτό και η συμβουλή που μπορώ να δώσω σε όλους και όλους εμάς είναι να κοιτάξουμε μέσα μας και μάλιστα με πολύ προσοχή διότι μπορεί κανείς να προσφέρει βοήθεια προς τα έξω, αλλά να κάνει και σχόλια προς τα έξω, μόνο όταν τα σχόλια αυτά που κάνει προς τα έξω τα κάνει και προς τα μέσα, προς τον εαυτό του. Και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό θα εξαρτηθεί, δηλαδή να είναι αξιόπιστη και προς τα μέσα. Στην αξιοπιστία αυτή συγκαταλέγεται επίσης και υποχρέωση τήρησης των υπεσχημένων και γι' αυτό λέω εδώ ρητά ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική συνεργασία με την Ουκρανία είναι κέρια σημασίας. Δεν μπορούμε να αρκούμαστε μονάχα σε υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Πρέπει αυτές να υλοποιηθούν. Ίσως εκεί θα πει περισσότερα ο Επίτροπος Χάν. Αυτό ισχύει και για πολύ δύσκολα και περίπλοκα θέματα όπως των προξενικών θεωρήσεων. Πάντως μπορείτε να υπολογίζετε στην εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης θερμά όλες και όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιτυχία της συνεργασίας Στην σύνταξη της εκθέσεως που έχει περιλάβει τις σκέψεις του Πατ Κόξ, ο οποίος θα μου την υποβάλει, σχετικά με μια συνέχεια. Δεν αρκεί να συνταχθεί μια ωραία έκθεση και μετά η έκθεση αυτή να καταλήξει στα συρτάρια. Γι' αυτό νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις του Πατ Κόξ. Εγώ προσωπικά θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων και το λέω καθαρά αν ο συνάδελφος Κόξ συνεχίσει να εργάζεται πάνω στην προσπάθεια υλοποίησης των συστάσεών του. Έχει τόσο πολύ εργαστεί πάνω στην υπόθεση αυτή που είναι σχεδόν πια Ουκρανό. Σας εύχομαι σε όλε και όλους καλή επιτυχία στην εργασία σας εδώ. Σας ευχαριστώ εγκαρδίως για την συνεργασία σας και σας διαβεβαιώ και πάλι και νομίζω πάντω στο όνομα της συντριπτικής πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας διαβεβαιώ ότι βρισκόμαστε στο πλευρό της χώρας σας που αντιμετωπίζει προκλήσεις παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, που αγωνίζεται για το μέλλον του και που χρειάζεται στήριξη, που την στήριξη αυτή μπορεί να την λάβει από εμάς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Thank you very much, President Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Σούλτς. Και τώρα ο λόγος αμέσως στον πρόεδρο Γκρόισμαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. με πρόεδρε Σούλτ, κύριε Μπρόκ, κύριε Πλένκοβιτς, με κύριε Κόξ, κύριε πίτρο Πεχάν. συνάδελφοι. Πρωτίστως και καταρχήν ήθελα να εκφράσω την ευχαριστίες μου για την ενίσχυση της συνεργασίας μου της συνεργασία μας και την ε, καλή σας διάθεση να λήξει η οποιαδήποτε σύγκρουση στην Ουκρανία. Ε, νομίζω ότι αυτή η στιγμή θα καταγραφεί στην ιστορία της Ευρώπης και της Ουκρανίας ως ημέρα που κηρύσσει την έναρξη της ποιοτική και τολμηρή αλλαγή στον νεοβουλευτισμό στην Ουκρανία ποτέ στο παρελθόν στην ε, σχέση μας με την Ευρώπη δεν είχαμε τέτοια παρουσία ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτό είναι και λογικό αλλά και συμβολικό ταυτόχρονα. Και εσείς αλλά και εμείς αντιμετωπίζουμε μια σωρία προβλημάτων στα οποία πρέπει να αντιδράσουμε με τον σωστό τρόπο. Οι σχέσεις μας έχουν πάρει λοιπόν μια τελείως διαφορετική χρειά. Ε, η συγκυρία της ε, συμφωνίας αυτής με το Μνημόνιο κατανόηση την παρουσία του, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουκρανία, την αποστολή για την ε, καταγραφή των αναγκών του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, και τις ανάγκες εξυγχρονισμού, εξυγχρονισμού του συγκεκριμένα. Όλα αυτά για μας είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες και σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα και να τα κάνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Σήμερα λοιπόν θέλουμε ακριβώ να ε, συζητήσουμε μαζί σα αυτέ τι αλλαγέ ώστε το Ουκρανικό Κοινοβούλιο να είναι ένα έμπροστο και διαφανή θεσμό. Να αρχίσει να έρχεται πιο κοντά στα πρότυπα των ευρωπαϊκών θεσμών. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι, όπω γνωρίζουν και όλοι, πόσο ε, ε, σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε τι δυσκολίε που περνάει από τη στιγμή η Ουκρανία λόγω εξωτερικών προκλήσεων και πιέσεων που οδηγούν, οδηγούν προκαλούν περισσότερη αστάθεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Η πολιτική κρίση την οποία περνάμε δεν είναι ανάγκη να χαρακτηρίζεται με όρους υπερβολικού, είναι μια κυβερνητική κρίση. Και σε κοινέ διαβουλεύσει και συζητήσει με την πλειοψηφία των βουλευτών στην Ουκρανία, ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλοι θέλουμε αποτελεσματικέ δραστικέ λύσει που δεν θα ανακόψουν την ευρωπαϊκή μα πορεία, αλλά θα ενισχύσουν τι ευκαιρίε που έχουμε στι σχέσει μα με την Ευρώπη. Θα ενισχύσουν του δημόσιου θεσμού μα και θα επιτρέψουν στην φίλη ευρωπαϊκή πλειοψηφία στη χώρα να περάσει τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε η κοινωνία μας να μεταλλαχθεί και να υπάρχουν σταθεροί μηχανισμοί για να προλάβουμε μελλοντικές κρίσεις. Ούτε πολιτικές, ούτε κοινωνικές, ούτε οικονομικές στο μέλλον. Αυτό είναι το καθήκον μας και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε ότι τα πάντα έχουν τελειώσει και ότι πρέπει να περάσουμε σε εκλογέ. Δεν είμαι βέβαιο ότι η πλειοψηφία όσων βρίσκονται εδώ στην αίθουσα θα συμφωνούσαν. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε πριν οργανώσουμε εκλογέ. Έχουμε πολλέ ευκαιρίε που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε προκειμένου η χώρα μα να πετύχει. Όσο και αν υπάρχουν εμπόδια, όσο και αν υπάρχουν προσκόμματα, θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση και ταυτόχρονα θα πρέπει να αγωνιστούμε ώστε η Ράντα να ε, ε, μετατραπεί σε ένα χώρο σταθερότητα. με ε, το κράτο δικαίου να πρετανεύει. Η ρωσική επιθετικότητα δεν είναι λόγο για να σταματήσουμε ή να καθυστερήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτή ακριβώς η να καθυστερησουμε τι μεταρρυθμισει αυτη ακριβω η αυτό που θα ήθελε η Μόσχα αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε να περάσει το δικό τους. Σήμερα λοιπόν η παρουσία μας εδώ δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση προς το Ευρωκοινοβούλιο στις σχέσεις του Ευρωκοινοβουλίου με την Βερχόφτα Ράντα της Ουκρανίας. Είναι ένα δείγμα ότι η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής και Ένωσης και Ουκρανίας προχωρά. Ότι οι σχέσεις μας είναι ουσιαστική και όχι απλώς στα λόγια. Η συμφωνία σύνδεσης βέβαια Ε, θα πρέπει να οδηγήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις όπως και η σχέση μας, αυτή η προνομιακή σχέση που έχουμε με το Ευρωκοινοβούλιο ως Ράντα. Θέλουμε να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ουκρανία. Ήδη από πέρσι νέα τεχνολογικά μέσα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε υπερχόφνα Ράντα προκειμένου να έχουμε καλύτερη διαχείριση και περισσότερη διαφάνεια των κυκλοφορικών εργασιών προ του πολίτε. Αλλά αυτή δεν είναι μόνο η μόνη αλλαγή. Είναι πολλέ οι αλλαγέ που οι Ουκρανοί βουλευτέ ε, καλούνται να πραγματοποιήσουν καθημερινά και υπάρχουν και πολλά προβλήματα που συνεχώ ε, προκύπτουν. Το θέμα λοιπόν είναι η προσέλευση, η συστηματική παρουσία, η δεοντολογία, η διαφάνεια συμφωνώ με όλα, όλες αυτές τις προτεραιότητες. Θα πρέπει ε, η διοικητική μας μηχανή να εξοπλιστεί καταλήλως. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να επανδρωθούν σωστά και ο υπερβολικό φόρτος εργασίας κάποιες φορές ε, για την ε, μελέτη των νομοσχεδίων είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν θέλουμε να αποδυναμωθούν ε, θεσμικώ ε, οι δομέ τη χώρα, ιδίω η Φερκόπνα Ράντα, και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προ την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Σούλτ και τον κύριο Πλένκοβιτ για τη στήριξη των προτάσεών μα, για να οργανωθεί και άλλη αποστολή προ την Ράντα για την αποτίμηση των αναγκών. Ευχαριστώ επίση όλου του απεσταλμένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, προθυμία του να συνεργαστούν μαζί μα και να ενισχύσουν στο έργο του τη Βερχόφνα Ράντα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη συνεργασία σα, κυρίε και κύριοι. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Κόξ για την ποιοτική και χωρί προκαταλήψει διάγνωσή του για το πώ λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Βερχόφνα Ράντα. Ε, χάρη στη δική του ηγεσία του τελευταίου μήνε μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε μια πολύ καλή καταγραφή τη πραγματικότητα. Θα ήθελα ξεκάθαρα να δηλώσω ότι η έκθεση που υποβάλλουμε σήμερα είναι μια έκθεση κοινή, μια κοινή καταγραφή της προσπάθειας των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου και της Ουκρανίας. Αυτή η κοινή ε, έμπνευση της έκθεσης επιτρέπει να καταρτήσουμε τις αδρές γραμμές και έναν οδικό χάρτη για το πώς θα προχωρήσουμε. Τι θα πρέπει να επιδιώξει η από πολιτική σκοπιάς και πώς θα μπορέσει να καλύψει τις προσδοκίες και τα συμφέροντα όλων των Ουκρανών πολιτών. Αυτή θα είναι η συνεισφορά μας σε ένα μέλλον σταθερότητας για την Ουκρανία. Ε, θέλουμε ένα ισχυρό θεσμικό όργανο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, να προβλέπει τους κατάλληλους κανόνες και νόμους και να είναι πρότυπο δημοκρατικής ε, λειτουργίας ασχέτως του ποιος προεδρεύει ή ποιος βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Θέλουμε αυτή η ιστορική μεταρρύθμιση να ολοκληρωθεί και να επικεντρωθεί στο γεγονό ότι δεν μα απασχολούν πλέον τα άτομα, αλλά οι θεσμοί, οι δομέ. Κάποια στιγμή η κρίση και οι απειλέ που αντιμετωπίζουμε δεν θα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στην Ουκρανία. Ελπίζω ότι η πλειοψηφία συμμερίζεται την άποψή μου θα πρέπει η φρύχοφνα Ράντα να είναι ένα κλειοδότημα που θα αφήσουμε στο μέλλον για να επιλύονται όλε οι μελλοντικέ κρίσει με έναν τρόπο σταθερό και προβλέψιμο. Ένα τέτοιο κοινοβούλιο, ισχυρό και ευρυθμό, θα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα ποιε κρίσει προκύψουν με τρόπο επαγγελματικό. Αυτή θα είναι η κοινή μα νίκη. Όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσει, λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μεταρρύθμιση ξεκινάει από εμά του ίδιου. Δηλαδή, η υλοποίηση αυτού του κοινού προγράμματο θα επιτρέψει ο κοινοβουλευτισμό στην Ουκρανία να έχει ένα νέο πρόσωπο. Αυτό ακριβώ μα ενδιαφέρει. Το κοινοβούλιο τη Ουκρανία ε, οφείλει να ξεκινήσει με μεταρρυθμίσει, να αναγεννήσει τι ε, δικέ του θεσμικέ δυνατότητε και όλη τη υπόλοιπη ε, δομή των δημόσιων αρχών στην Ουκρανία. Μαζί για μια κοινή νίκη λοιπόν. Σα ευχαριστώ πολύ. Äh, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο λαμβάνει ο πρόεδρος Πατ Κόξ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Φερχοφναράντα, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε Μπροκ, κύριε Πλένκοβιτς, κύριε Τομπίνσκι, πρέσβη του Τομπίνσκι, ε, αξιότιμοι καλεσμένοι. Για μένα είναι μια στιγμή συγκίνησης αυτή. Βλέπω τόσου ανθρώπου συγκεντρωμένους σε αυτό το χώρο την ίδια στιγμή για να μοιραστούμε όλοι, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί, την αποφασιστικότητα και την διάθεση να πράξουμε και να ενεργήσουμε από κοινού για τα κοινά μα, τα συλλογικά μα συμφέροντα. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο και την Περχόφνα Ράντα που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μοναδική. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Πλέγκοβιτ, τον κύριο Μπροκ και όλου του συναδέλφου που ανέλαβαν ε, την ε, ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Δεν θέλω να θεωρηθώ εγώ ως ε, ο υπεύθυνο και ο εμπνευστή της έκθεση αυτής γιατί είναι ομαδική. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλη την ομάδα συνεργατών του Ευρωκοινοβουλίου για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους καθώς και τους συμβούλους μας διεθνώς και από την Ουκρανία που ε, μπόρεσαν με τον επαγγελματισμό τους να επιτρέψουν τη σύνταξη αυτού του εγγράφου. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τους διεθνείς μας εταίρους, καθώς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που μας ε, διευκόλυναν στην όλη μας προσπάθεια. Ιδιαιτέρως ευχαριστίες για τον πρόεδρο Γκόισμαν, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τους αντιπροέδρους, τους ε, Προέδρους Επιτροπών και τους βουλευτές. Όλοι μας έδωσαν τη δική τους οπτική γωνία και πολλά, πολλοί από τους βουλευτές ε, ή από τα μέλη της διοίκησης της Ράντα τους ευχαριστούμε που άνοιξαν τις πόρτες των γραφείων τους και ε, άφησαν την αποστολή μας να λάβει γνώση όσων πληροφοριών ήταν απαραίτητες. Γνώρισα ανθρώπους άξιους. Κάποιοι από εκείνους εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε αυτές τις προποθέσεις και τους όρους υπό τους οποίους εργάζονται. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν να πετύχουν το καλύτερο για τη χώρα τους. Ισχύει παντού αυτό. Τα πολιτικά πράγματα και οι ισχυρές προσωπικότητες πάνε μαζί. Επίσης, ε, πάλι ισχύει παντού ότι ο πρώην σοβιετικός χώρος σημαίνει ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες που συνυπάρχουν με αδύναμους πολιτικούς θεσμούς. Εάν υπάρχει μία φιλοσοφία που έχει εμπνεύσει όλη λοιπόν αυτή την έκθεση, είναι η πεποίθηση ότι η λύση για την μεταμόρφωση της δημοκρατίας, της κοινωνίας, της οικονομίας και του συστήματος δικαιοσύνης στην Ουκρανία είναι να χτίσουμε ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς. Ο Ζαν Μονέ ήταν εκείνος που ενέπνευσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την προσπάθεια, τη διαδικασία ένωσης της Ευρώπης και θα σας πω τα λόγια του έλεγε ότι τίποτα δεν είναι ε, δυνατό να συμβεί αν δεν βοηθήσουν οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες. Αυτό είπε τότε. Αλλά επίσης είπε τίποτε δεν διαρκεί χωρίς θεσμούς. Και αυτό είναι μια βασική ε, συνταγή για να μπορέσει κανείς να έχει πρόοδο. Έχει πληγεί κέρια η Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Το αίμα των αθώων αποχήθηκε στην πλατεία Μαϊντάν κατά την επανάσταση αξιοπρέπεια στη χώρα. Το αίμα των αθών και τραυματισμένων στον Ταμπάζ είναι τέτοια τραύματα. Ένας μεγάλος ε, φιλόσοφος του διαφωτισμού που ήταν καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Ιδιμβούργου, David Hume, έλεγε ότι όταν αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε, η πραγματική θεραπεία αρχίζει τότε. Τότε όταν υδρώνουμε και δεν χύνουμε αίμα, τότε αρχίζει πραγματικά η επούλωση. Αυτό λοιπόν προς τον πρόεδρο Γκρόισμαν, τους αντιπροέδρους και τους προέδρους των κομμάτων, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τους συνεργάτες μας από διεθνείς οργανώσεις στην Ουκρανία που προσπάθησαν για αυτή την μεταρρύθμιση, πρέπει να πω ότι είναι πεποίθησή μου, σταθερή πεποίθηση, ότι η διαδικασία μεταμόρφωσης και αλλαγής θα υλοποιηθεί όταν όλοι μαζί ιδρώσουμε με τον ιδρώτα του μετόπου μας, δουλέψουμε ε, για τη νέα Ουκρανία. Για μια νέα Ουκρανία των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των βουλευτών, των μελών της κυβέρνησης και όλων. Και να πω ότι πολλά από τα συμφέροντα που μπορεί να είναι κρυφά ή να αποκαλύπτονται ε, μπορούν με μία φράση να καλυφθούν. Κάποτε στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο του 1961 υπόθηκε από τον νερό πρόεδρο Κένεδη που ε, εκφώνησε μια ομιλία και είπε κάτι στους Αμερικανούς που θα το έλεγα και εγώ σήμερα στους ε, Ουκρανούς. Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει για σας η χώρα σας, αλλά ως Ουκρανοί ρωτήστε εσείς τι μπορεί να κάνετε για τη δική σας χώρα η έκθεση που έχετε μπροστά σας είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ήθελα να σας πω ότι χθε και σήμερα συνάντησα τους ηγέτες της Φερκοπναράντα και πραγματικά αναθάρισα. Αναθάρισα από το πόσο ενωμένοι είστε σε ένα κοινό σκοπό. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς όλους σας. Αυτήν την ενότητα αυτή την αλληλεγγύη, την ομοψυχή που την εκφράσατε στις Βρυξέλλες, να την ξαναπάτε στο Κίεβο. Και με το ίδιο πνεύμα ιδρώνοντας όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό, να πετύχετε, να πετύχετε στην οικοδόμηση μια νέας Ουκρανίας. Ο καθένας θα λάβει ένα αντίτυπο της έκθεσης αυτής μετά την ολοκλήρωση αυτής της ε, τελετής και η έκθεση θα διατεθεί και επιγραμμικά στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου, από απόψε στα αγγλικά και στα ουκρανικά. Και από την πλευρά της αποστολής παρατήρησης αναγκών είναι το δικό μου ευχάριστο καθήκον να υποβάλλω το αντίτυπο στα ε, ουκρανικά στον ε, πρόεδρο Γκρόσμαν και στα αγγλικά στον πρόεδρο Σούλτς το απάβγασμα της συλλογικής μας εμπειρίας για το ε, λαμπρό ελπίζω μέλλον σας. Dank, Pet. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο λαμβάνει τώρα ο Επίτροπος κύριος Χάν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εσείς οι υπόλοιποι κύριοι Πρόεδροι. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συνεργάτες του για την διοργάνωση της εβδομάδας Ουκρανίας καθώς επίσης και για την έλευση των Ουκρανών βουλευτών εδώ στις Βρυξέλλες σε μια δύσκολη περίοδο, τα εξήγησε αυτά ο πρόεδρος Σούλτς, θα σκεφτόταν ίσως κανείς ότι έχουμε και άλλα πιο σημαντικά να κάνουμε. Όχι, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο διάλογος και η συνεργασία και να δοθεί ένα θετικό παράδειγμα και εντός και εκτός Ευρώπης. Ότι είναι δηλαδή δυνατόν να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή και να εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι όλες και όλοι επιθυμούμε επιτυχία και ευχόμαστε επιτυχία στην Ουκρανία από την ε, άποψη, από τη σκοπιά της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλήρης υποστήριξη και για την διατήρηση της εδαφικής ακερότητας της χώρας σας. Δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό εδάφους. Θα πρέπει να εφαρμοστούν τα πράγματα ως έχουν συμφωνηθεί και μόνον τότε όταν έχει εφαρμοστεί η συμφωνία στο σύνολό της θα μπορέσουν να αρθούν οι κυρώσεις. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία και το γνωρίζουμε αυτό απολύτως καλά. Αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως πρόφαση για να καθυστερήσουν οι πολύ αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή. Ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες λόγω του μεγέθους της χώρας και του αριθμού των καθήκον της. Έχοντας γνώση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ουκρανία και που πιθανότατα είναι και μοναδικές ανά τον κόσμο επί του παρόντος, παρόλα αυτά οφείλει να γνωρίσει κανείς ότι επιτεύχθηκαν και σημαντικά βήματα προόδου τον προηγούμενο χρόνο και αυτά οφείλονται ασφαλώς στην εργασία και στη συνεργασία σας. Η προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας. Είναι κλασικό βήμα προς τα εμπρός. Άκουσα πρόσφατα ότι αυτό το ουκρανικό κρασί που έχει και θαυμάσια γεύση το βρίσκει πλέον κανείς και σε καταστήματα των Βρυξελών και όχι μόνο σε υπερκαταστήματα, σε σούπερ μάρκετ δηλαδή και σας καλώ να ψάξετε να το βρείτε και να το γευθείτε Σίγουρα και άλλες ε, σπεσιαλιτέ της χώρας αυτής θα βρούμε σύντομα στα καταστήματα, είμαι βέβαιος. Όμως υπήρξε σημαντικός αριθμός βημάτων πρόοδου, το είπα αυτό. Υπάρχουν και πολλά ανοιχτά πράγματα ακόμα. Σε ό,τι αφορά ας πούμε την ικανότητα του νομοθετήν, ας το πω έτσι. Καλά τα πάει η Ουκρανία. Αυτό που λείπει είναι η αιμονή στην εφαρμογή των νομοθετικών αποφάσεων και η βιωσιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και μιλώ για την μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, για την καταπολέμηση πραγματικά σε βάθος και σε πλάτος της διαφθοράς και εντός Ουκρανίας και εκτός Ουκρανίας συνομιλώ με εκπροσώπους επιχειρήσεων και ρωτώ τι γίνεται με την διάθεσή σας να επενδύσετε στην Ουκρανία και μπορώ να σας μεταφέρω τις απόψεις τους ότι δηλαδή συνολικά καταρχήν θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα επί το θετικότερο υπάρχουν όμως πολλοί ακόμη που διστάζουν να επενδύσουν ακριβώς λόγω των σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς και τοπικά και περιφερειακά. Για παράδειγμα, για την απόκτηση οικοδομικών αδειών, για την απόκτηση αδειών λειτουργία εργοστασίων και Αυτά είναι κρίσιμα πράγματα και πρέπει να συζητηθούν. Εδώ τίθεται και το θέμα της απελευθέρωσης των προξενικών θεωρήσεων. Γνωρίζω ότι αυτό σας απασχολεί πολύ και σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τα πράγματα. Αλλά για να είμαι και ειλικρινής, από εσά εξαρτάται εν, τέλει, δηλαδή και από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, εάν θα λάβετε τις σχετικές αποφάσεις με τέτοιον τρόπο που να σέβονται και να συμμορφώνονται τα ήδη διατυπωθέντα κριτήρια. Για παράδειγμα, της ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και των βουλευτών της Ράντα. Εκεί υπάρχει ακόμα ανάγκη να γίνουν κάποια πράγματα, διότι είναι αναγκαίο να είναι ξεκάθαρα τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών και τώρα βεβαίως, αλλά και ε, στρέφοντας τα βλέμματα προς το παρελθόν και όχι μόνο προς το μέλλον. Πάντως είναι πράγματα τα οποία εάν υπάρχει η πολιτική βούληση μπορούν να προωθηθούν γρήγορα και να εφαρμοστούν γρήγορα. Υπό το πνεύμα αυτό επιθυμώ να σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες σας που είμαι βέβαιος ότι το έργο σας δεν είναι καθόλου εύκολο. Η Ουκρανική Βουλή έχει και ένα χαρακτήρα υποδείγματος και για τις βουλές άλλων γειτονικών χωρών και αποτελεί πραγματικό παράδειγμα διότι και σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή σας αλλά και διότι φέρετε ακόμα μέσα σας το πνεύμα της πλατείας του Μαϊντάν. Και έτσι έχετε, εμπνέεστε από αυτή την υψηλή ηθική υποχρέωση και η χρονομία. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε συγκεκριμένα κόμματα υποστηρίζουμε, ούτε μονομένα άτομα. Εμείς στηρίζουμε αρχές, την πολυφωνία, την διαφάνεια, την δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Αυτά είναι τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Ουκρανία είναι μέρος της Ευρώπης και έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Ουκρανία να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο την Ευρώπη. Και στο πνεύμα αυτό, ξαναλέω, σας καλώ να συνεχίσετε το έργο που έχετε αναλάβει και αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο σχόλιο, είναι αναγκαίο νομίζω να το επισημάνω αυτό, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία του ότι δεν αντιμετωπίζετε εκλογές για τα μέσα επόμενα χρόνια. Ρίξτε το βάρος σας στην εφαρμογή των συμφωνημένων η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν την διάθεση και την θέληση να συνεργαστούν μαζί σας. Αλλά πρωτίστως αυτό, η προσπάθεια αυτή πρέπει να ξεκινά από εσά. Αυτό αναμένουν άλλωστε και οι Ουκρανοί από εσά. Και όπως είπε και ο πρόεδρος Σούλτς, το τονίζω και εγώ, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα προόδου, στο μέλλον θα είναι δεδομένη η οικονομική στήριξη. Και θα έλεγα μάλιστα όχι μόνο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και των διεθνών πιστοτικών οργανισμών. Διότι όλοι έχουν ενδιαφέρον η Ουκρανία να αποδειχτεί ιστορία επιτυχίας και να δείξει έτσι το καλύτερο παράδειγμα ότι μια ειρηνική στραμμένη προς το μέλλον συνεργασία βασισμένη στη δημοκρατία μπορεί να ξεπεράσει τα κολλήματα που επιβάλλει το παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στρέφω τα βλέμματα στην αίθουσα, βλέπω πολλά γνωστά πρόσωπα και από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό. Ήδη από τότε, από το 2004-2005, το Μαϊντάν 1, μετά μας ήρθε το Μαϊντάν 2 και ελπίζω ότι μάθαμε κάτι από τα διδάγματα του Μαϊντάν 1 και ότι τώρα θα μπορέσουμε στη βάση αυτών των συμπερασμάτων να προχωρήσουμε σε νέα βήματα. Δημοσκοπήσεις που μπορεί να καταγράφουν τις αλλαγές της απόψεις των ψηφοφόρων δεν μπορούν να αποτελούν την βάση για την πρόκληση εκλογών. Χρειάζεται σταθερότητα, ηρεμία για τα επόμενα χρόνια για να προχωρήσει το νομοθετικό έργο. Σας εύχομαι ευχάριστη διαμονή. Στις 6 το απόγευμα προβλέπεται δεξίωση και από αύριο θα στρωθούμε στη δουλειά. Σας ευχαριστώ.